Colleagues, does the microphone actually work? Ε, συνάδελφοι, ακούτε, με ακούτε, δουλεύει το μικρόφωνο. I don't hear very much. Γιατί δεν το ακούω καλά. Can you try again? Hello? Yeah, this sounds better. Yes, thanks. Okay, good afternoon. Good... Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε αυτήν την ε, συνεδρίαση τη... της Ανακριτικής Επιτροπής. μάλλον πλησιάζουμε σε αυτή, έχουμε ακόμα μερικές συνεδρίες. Πριν να σας πω το σημερινό πρόγραμμα, θα ήθελα να χαιρετήσω τους επισκέπτες της κυρίας Μορφάη, όλες γυναίκες μάλλον. Γεια σας. Συνάδελφοι, σήμερα θα μιλήσουμε, δεν θα γίνει η παρουσίαση για τους μηχανισμούς παρακολούθησης του Γερμανικού Κοινοβουλίου, γιατί τώρα γίνεται η νέα κυβέρνηση συνασπισμού και η παρουσίαση του εγγράφου εργασίας των κυρίων Μωράης και Κίρκχοπε για το πεδίο της διεθνούς ευρωπαϊκής και εθνικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και αυτό αναβάλλεται για μια άλλη συνεδρίαση. Εάν λοιπόν συμφωνείτε, εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη με αυτές τις ε, αλλαγές. Ωραία, δεν υπάρχει αντίρρηση. Σήμερα έχουμε δύο συνεδρίες. Η μία για την παρακολούθηση των ε, μυστικών υπηρεσιών σε εθνικό ε, επίπεδο, σε μια εποχή μαζικής ε, παρακολούθησης. Θα ακούσουμε τον κύριο Μίκαλ Τέτσνερ, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Παρακολούθησης και Συνταγματικών Υποθέσεων της Νορβηγίας και από τις 4 και μετά θα έχουμε την παρουσίαση του εγγράφου εργασίας για τις δραστηριότητες παρακολουθήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά τα ευρωπαϊκά δεδομένα και τις πιθανές νομικές ε, επιπλοκές για τις υφιστάμενες ε, διατλαντικές συμφωνίες και τη συνεργασία. Οι εισηγητές είναι και συγγραφείς ο κύριος Μωράης και Βος και θα σταματήσουμε στις 5. Από ό,τι βλέπω, δεν έχουμε πολλούς ε, ευρωβουλευτές εδώ παρόντες. Ε, θα ήθελα όμως παρόλα αυτά να σας ζητήσω να είστε συνοπτικοί στις ερωτήσεις και στις απαντήσεις σας και αν υπάρχει ανάγκη θα κάνουμε και ένα δεύτερο γύρο. Με χαρά μου λοιπόν καλωσορίζω τον κύριο Μάγκλ Τάτσνερ σας δίνω το λόγο για μια σύντομη παρουσίαση των μηχανισμών παρακολούθησης στην Νορβηγία και μετά ανοίγει ο διάλογος. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Η Νορβηγία δεν είναι ακόμη επίσημη γλώσσα της, ε, ε, ε, επίσημη, επίσημος, δεν έχει ακόμα επισήμως αναγνωριστεί η νορβηγική γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω τα δανέζικα στην παρουσίαση. Εάν δεν σας πειράζει, λοιπόν, είμαι έτοιμος. Καταρχάς, ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου αποστήλατε που μας αποστήλατε για να έρθω εδώ να σας συναντήσω και να σας παρουσιάσω την ε, λειτουργία του Νορβηγικού Κοινοβουλίου σχετικά με τις μυστικές υπηρεσίες. αυτό το... Αυτή η δραστηριότητα, ε, η δραστηριότητα του ελέγχου μάλλον, είναι ε, μία από τις βασικές του Κοινοβουλίου μας. Αυτό σημαίνει ότι η κυβερνητική πολιτική βασίζεται στις κοινοβουλευτικές πράξεις. Έχουμε 12 κοινοβουλευτικές επιτροπές στο Νορβηγικό Κοινοβούλιο και ο έλεγχος είναι πολύ σημαντικός. Ε, πρόκειται ε, για την Επιτροπή Ελέγχου και Συνταγματικών Υποθέσεων που αναλαμβάνει αυτή, ε, αυτό το εγχείρημα. Επίσης έχουμε και τέσσερους εξωτερικούς που εκ μέρους του Κοινοβουλίου αναλαμβάνουν τον έλεγχο. Είναι για παράδειγμα το ελεγκτικό συνέδριο, διαμεσολαβητής για τη δημόσια διοίκηση και ο διαμεσολαβητής για την άμυνα. Το, η τέταρτη επιτροπή είναι η EOS όπως ονομάζεται. Ε, αυτό είναι το νορβηγικό ακρόνιμο ακρονίμιο και αυτό θα είναι και το θέμα της παρουσίασής μας. Είναι EOS σημαίνει ε, υπηρεσία ε, προστασίας ε, εσωτερικής ασφάλειας ε, και μυστικών υπηρεσιών. Πρόκειται για μια ειδική πράξη του Κοινοβουλίου, η οποία ίδρυσε αυτή την Επιτροπή. Το, υπόβραθ, το υπόβαθρο για τη δημιουργία αυτή της Επιτροπής ήταν ένας ε, ευρύς δημόσιος διάλογος σχετικά με τις δραστηριότητες των μυστικών υπηρεσιών στην Νορβηγία. Υπήρξε μεγάλη κριτική το 1994 το Κοινοβούλιο δημιούργησε λοιπόν μια επιτροπή για να εξετάσει τις υπηρεσίες, τις μυστικές υπηρεσίες. Η έκθεση αυτής της ε, επιτροπής ε, είχε ως ε, συμπέρασμα ότι οι εποπτικές υπηρεσίες, ειδικότερα στην δεκαετία του 60 και του 70, ε, είχαν παρακολουθήσει ε, σε πολιτικό επίπεδο ε, πολλά άτομα. Γενικά <clears throat> ήταν εκτεταμένη αυτή η παρακολούθηση. Ένας από τους όρους, μία από τις πηγές αυτής της συζήτησης και ένα από τα αποτελέσματά της ήταν αυτή η δημιουργία της Επιτροπής EOS. Όσον αφορά λοιπόν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ξεκίνησε με αυτήν την ε, αφετηρία. Η Επιτροπή ΟΕΣ είναι μόνιμη Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Τα μέλη επιλέγονται από το Κοινοβούλιο για μια θητεία 5 ετών. Υπάρχουν 7 μέλη και προσπαθούμε τα μισά μέλη μας ε, περίπου να είναι πολιτικοί. Συχνά είναι και πρώην μέλη του Κοινοβουλίου, ενώ το άλλο κομμάτι της Επιτροπής αποτελεί, ε, αποτελείται από πρώην ε, δικαστές, ερευνητές κτλ. Είναι η νορβηγική κοινωνία των πολιτών που εκπροσωπείται. Υπάρχει επίσης και η γραμματεία από δικηγόρους απαρτίζεται και τα μέλη της έχουν ε, δυνατότητα πρόσβασης, μέγιστη δυνατότητα πρόσβασης. Βέβαια πάντοτε υπόκεινται στους όρους της εμπιστευτικότητας. Ο βασικός ε, σκοπός αυτής της ειδική Επιτροπής είναι η διασφάλιση της, ε, και της προστασίας των πολιτών. Η προστασία των πολιτών έναντι των ε, εποπτικών υπηρεσιών. Θέλουμε να προστατέψουμε τα δικαιώματα των πολιτών έναντι των υπηρεσιών αυτών, έτσι ώστε να μην βλάπτουν οι υπηρεσίες αυτές την πολιτική ζωή στην Νορβηγία. Πέρα από αυτό το στόχο, προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε και την συμμόρφωση με την νομοθεσία. Πρόκειται για έναν γενικότερο έλεγχο. Δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Το κριτήριο είναι ότι αν μία κρατική υπηρεσία ασχολείται με την ε, παρακολούθηση, την εποπτεία και την ασφάλεια, υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Το μεγαλύτερο μέρος του ελέγχου έχει να κάνει με τις παραδοσιακές μυστικές υπηρεσίες, όπως ε, για παράδειγμα αυτές της αστυνομίας και του στρατού. Η Επιτροπή έχει το ελεύθερο να ελέγχει. Υπάρχουν επιθεωρήσεις, περίπου 30 το χρόνο γίνονται, 30 περίπου τέτοιοι έλεγχοι. Και δεύτερον έχουμε και παράπονα πολιτών που λαμβάνουμε γύρω στα 30 ε, κάθε χρόνο. Η Επιτροπή λοιπόν αρχίζει η διαρεύνηση των παραπώνων αυτών και να πω επίσης ότι έχει και σχεδόν απεριόριστα δικαιώματα ελέγχου. Έχει πρόσβαση σε όλα τα αρχεία και τα μητρώα. Επίσης έχει πρόσβαση σε όλα τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις. Μπορεί επίσης να καλέσει τις υπηρεσίες και τη διοίκηση για να εξηγήσουν τι ακριβώς κάνουν πάντοτε βάσει των κανόνων που χρησιμοποιούνται για την εξέταση των μαρτύρων στα δικαστήρια. Υπάρχει ένα πλαίσιο για αυτούς τους ελέγχους, για αυτές τις επιθεωρήσεις. Ο έλεγχος της αστυνομίας είναι τουλάχιστον έξι φορέ το χρόνο, ενώ στο στρατό ο έλεγχο των μυστικών υπηρεσιών γίνεται τουλάχιστον δύο φορέ το χρόνο. Πέρα από αυτό υπάρχουν και οι περιφερειακές οργανώσεις των υπηρεσιών εκείνων που ελέγχονται. Κατά κανόνα ε, θα πρέπει να ανακοινώνονται εκ των προτέρων οι έλεγχοι, όμως υπάρχει δυνατότητα και ευνίδιων ελέγχων. Και αυτό συμβαίνει συχνά, θα έλεγα. Αν κάποιος πολίτης θεωρεί ότι ότι μία από τις ε, υπηρεσίες ασφάλειας, οι μυστικές υπηρεσίες, ε, ε, τον έχει βλάψει κατά κάποιο τρόπο, τότε γίνεται μία έρευνα. Τα παράπονα συνήθως έχουν να κάνουν με κριτική των υπηρεσιών. Όπως είπα όμως προηγουμένως, υπάρχουν και κατά πρωτοβουλία ε, έλεγχοι που γίνονται από το Κοινοβούλιο. Και ως αποτέλεσμα αυτών ε, βγαίνουν κάποιες ε, εκθέσεις. Για την αστυνομία, για παράδειγμα, η Επιτροπή θεώρησε ότι η νομιμότητα των μεθόδων πρέπει να αξιολογείται πριν από την ούτως αποκαλούμενη υπόθεση Τρίχολτ η αστυνομία είχε τη δυνατότητα να ακούει ας πούμε τις τηλεφωνικές ε, συνδιαλέξεις κάποιου, αλλά όχι αυτά που συμβαίνουν μέσα στο σπίτι τους, τα δωμάτια. Μετά είχαμε την αστυνομική καταχώρηση δύο Ισλαμικών ομάδων. Αυτό ήταν μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Η Επιτροπή εξέτασε το πώς ε, αντιμετωπίζονται οι πολιτικές και θρησκευτικές απόψεις ε, στα μητρώα της αστυνομίας. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, βρέθηκε ότι η αστυνομία πήγε πέρα από τα όρια. Η τρίτη έκθεση είχε να κάνει με την παρακολούθηση και καταχώρηση Νορβηγών πολιτών που περνούσαν από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Νορβηγία, στο Όσλο. Η αστυνομία επικρίθηκε γιατί ε, δεν είχε σωστή πληροφόρηση για το σύστημα ασφάλειας μπροστά στην πρεσβεία και δεν υπήρχε και επικοινωνία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή υπάρχουν δύο υποθέσεις που εξετάζονται. Η μία έχει να κάνει με πληροφοριοδότες ε, της αστυνομίας ε, που έχουν διεισδύσει στην άκρα αριστερά. Και αυτό βγήκε σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Η Επιτροπή και τα ξεταρχία της ε, αστυνομίας έχει κάνει συνεντεύξεις, έχει ανακρίνει την, το προσωπικό της αστυνομίας και προχωρά την υπόθεση. Επίσης, για τις μυστικές υπηρεσίες βλέπει ότι δεν ακολουθούνται οι κανόνες και έγιναν και δύο εθνίδιοι έλεγχοι λόγω παραπώνων των πολιτών. Τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή επίσης έχει θεσπίσει και συνεργασία με άλλες ελεγκτικές επιτροπές, όπως αυτές της Σουηδίας, της Ολλανδίας και του Καναδά που είναι παρόμοιες με την δική μας επιτροπή, την EOS. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ελέγξει κανείς τις υπηρεσίες ασφαλείας. Ανεξάρτητα από τα μοντέλα που επιλέγεις, υπάρχει όμως ένας κοινός στόχος. Εργάζεσαι εκ μέρους των πολιτών και των ε, νομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους που πρέπει να γίνονται σεβαστά από τις ε, υπηρεσίες ασφαλείας. Οι υπηρεσίες ασφαλείας συνεργάζονται για την πάταξη της τρομοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει και έλεγχος ε, της σχέσης μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών ασφαλείας, δηλαδή της Νορβηγικής και αυτή, αυτών ε, των υπηρεσιών που ανήκουν σε άλλες χώρες. Έτσι λοιπόν οι ηλεκτρονικές ε, υπηρεσίες και οι πληροφορίες συγγνώμη, και τα ε, αναγκαστικά μέτρα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να ελέγχονται. Πρέπει να βρούμε δηλαδή τη χρυσή τομή μεταξύ των δικαιωμάτων των πολιτών και της ανάγκης για προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Υπάρχει υποστήριξη γι' αυτό μέσα στο στο ευρύ κοινό. Οι μέθοδοι όμως που χρησιμοποιούνται πολλές φορές είναι αμφισβητούμενες γιατί αυτοί που παρακολουθούνται πολλές φορές δεν το γνωρίζουν και ο στόχος αυτής της Επιτροπής είναι να αξιολογηθεί κατά πόσο αυτές οι μέθοδοι δεν ε, βλάπτουν στην ουσία τους ε, πολίτες, τα άτομα. Αυτή η αρχή λοιπόν είναι ε, πάγια, ότι η Επιτροπή πρέπει, πρέπει να διασφαλίζει όλα αυτά και να αναφέρεται στο Κοινοβούλιο. Το δίλημα του Κοινοβουλίου είναι το εξής. Ε, πρέπει να υπάρχει το απόρριτο σε αυτή την Επιτροπή, καθώς ε, ασχολούνται με απόρριτες πληροφορίες, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πέρα από το να πιστέψουμε αυτά που μας ε, λέει η Επιτροπή. Γίνεται μια ετήσια έκθεση ε, η οποία κατατίθεται στην Επιτροπή Ελέγχου και Συνταγματικών Υποθέσεων, στην οποία είμαι και μέλος και υπάρχει και εκεί η σύνταξη ενός ε, ψηφίσματος για το Κοινοβούλιο, στο οποίο συμμετάσχουν και οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Άμυνας. Υπάρχει λοιπόν ε, πολύ χώρος για να συζητηθεί ε, η δραστηριότητα, η αιτήσια δραστηριότητα των μυστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλείας. Υπάρχει συνένεση στην ε, Νορβηγία σχετικά με το, την ανάγκη για δημοκρατικό έλεγχο των υπηρεσιών αυτό έτσι ώστε να προστατέψουμε τη δημοκρατία. Η Επιτροπή Ελέγχου επιλέγεται από το Κοινοβούλιο και αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι επιτυχία. Ο στόχος της Επιτροπής είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Πρέπει ενεργά να αντιμετωπίζουν υποθέσεις μέσα στα πλαίσια της θητείας τους και οι ελεγκτικές τους δραστηριότητες είναι μεγάλη, ε, μεγάλη σημασία και συνεισφέρουν τα μάλα στην ε, δημοκρατία και στην δημιουργία της εμπιστοσύνης του λαού απέναντι σε αυτές τις υπηρεσίες. Ευχαριστούμε πολύ. Okay, thank you very much for the very interesting presentation. Um, I'll start with the shadow rapporteurs present, and then the first one on this would be Mr. Voss on behalf of the EPP. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Präsidentin. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω και εσάς για την ε, παρουσίασή σας. Έχω διάφορες Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για την παρουσίασή σας αυτή. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κύριε Τέτσνερ. Έχω διάφορες μικρές ερωτήσεις να σας κάνω. Καταρχάς, αυτά που μας ε, αναφέρεται έχουν να κάνουν με την ε, εσωτερική μυστική υπηρεσία. Υπάρχει κάποια εξωτερική μυστική υπηρεσία σε ό,τι αφορά την Νορβηγία, δηλαδή σε ό,τι αφορά την προστασία των νορβηγικών ε, ε, αρχών. Αυτό περιλαμβάνει τμήμα της, των εργασιών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής σας. Ύστερα, σε ό,τι αφορά τις μεμονωμένες περιπτώσεις, ήθελα να ρωτήσω, αυτές οι πληροφορίες για τα μεμονωμένα μέσα που λαμβάνετε, πόσο λεπτομερείς είναι. Είναι γενικής φύσεως, είναι πιο εξειδικευμένες. Ύστερα, θα με ενδιαφέρει να ακούσω από την περίπτωση, από την υπόθεση Μπράιβικ, έχει αλλάξει κάτι στη δομή και στα καθήκοντα που διαμορφώνονται των υπηρεσιών και της Επιτροπής. Επιπλέον, είπατε ότι όταν υπάρχουν καταγγελίες από τους πολίτες ε, συνεδριάζεται ε, υπάρχει και κάποια, κάποιο είδους ε, κατάσταση απειλητική κατεπίγουσης ανάγκης κατά την οποία συνεδριάζεται ή μόνο σε περίπτωση καταγγελίων. Και επίσης είναι μόνο οι Νορβηγοί πολίτες αυτοί που μπορούν να απευθυνθούν στην Επιτροπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σάψνερ. Ναι. Δεν κατάλαβα. Α, συγγνώμη, άκουγα τα γερμανικά. Ε, τα γερμανικά δεν άκουγα στην ε, γλώσσα τη επιλογή μου. Καταλαβαίνω όμω ε, λίγα γερμανικά να απαντήσω όμω με μια επιφύλαξη. Καταρχά, με ρωτήσατε κατά πόσο ο έλεγχος έχει να κάνει και με τις αλλοδαπές ε, ε, υπηρεσίες, ε, μυστικές υπηρεσίες της Νορβηγίας σε ό,τι αφορά το Αφγανιστάν για παράδειγμα. Ναι, όντως αυτό σημαίνει. Η Επιτροπή αυτή είναι αρμόδια για όλα, όλες τις υπηρεσίες ασφαλείας. Είτε μιλάμε για παρακολούθηση νορβηγών στο εσωτερικό της χώρας, είτε στην Ελλοδαπή. Δεν πιστεύω όμως ότι ε, έχουμε οποιαδήποτε δικαιοδοσία σε μη Νορβηγούς στο εξωτερικό. Πρέπει να υπάρχει κάποια σύνδεση με την Νορβηγία σε κάθε περίπτωση. Κατά δεύτερον, σε ποιο βαθμό μπορούμε να αξιολογήσουμε τις μεθόδους πολύ ενταλεχώς να σας απαντήσω σε ό,τι αφορά δηλαδή τις μεθόδους που εφαρμόζονται από τις μυστικές υπηρεσίες και σε ό,τι αφορά τα δηλαδή, θέματα ασφάλειας. Τα μέλη τώρα της Επιτροπής έχουν ε, έχουν τη μέγιστη άδεια το ελεύθερο να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες ό,τι αφορά και την ε, πρόσβασή του στο Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά δηλαδή τις μυστικές απόρριτες πληροφορίες. Όχι σε ονόματα κλπ. Αν το Κοινοβούλιο λοιπόν πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στην αξιολόγησή μα. προκειμένου να, έχουμε, να έχει και μια εντύπωση για το τι λαμβάνει η χώρα στο πλαίσιο των μυστικών αυτών υπηρεσιών. Κατά τρίτον, η τρομοκρατική επίθεση κατά των ε, πολιτών από τον Νορβηγό κύριο Μπράιβικ. Σε δύο τομείς πρέπει να σας πω ότι ασκήθηκε κριτική κατά των υπηρεσιών των αστυνομικών. Δεν ήταν αρκετά προσεκτικοί, δεν επέτυξαν τον απαραίτητο ζήλο. Ο δε επικεφαλής ε, των μυστικών υπηρεσιών της αστυνομίας τότε είπε, τότε δήλωσε ότι δεν ήταν δυνατή ο εντοπισμό ε, του κυρίου Βέβικ στο ραντάρ το αστυνομικό. Δεν υπήρχε δυνατότητα πλέον να υπάρχει ένα σύστημα τύπου στάζι. Και σε αυτό έχει ασκηθεί έντονη κριτική. Ναι, μεν δεν θέλουμε μια κοινωνία παρακολούθηση από την αστυνομία, από την άλλη όμω, σε συγκεκριμένη περίπτωση, στην συγκεκριμένη υπόθεση, οι αστυνομικέ υπηρεσίε καταφανώς δεν ε, αντιλήφθηκαν το επίπεδο του κινδύνου. Είχε εισαγάγει υλικά ο κύριος Μπράιβνικ για να κατασκευάσει μια μεγάλη βόμβα με τα αποτελέσματα που είδαμε. Μιλάω για τη μομιστική του επίθεση στα κτίρια τα κυβερνητικά. Αυτό ήταν το πρώτο τμήμα της επίθεσης. Το δεύτερο τμήμα ήταν η επίθεση κατά τον, ε, στο, στο νησί στο, κατά της ε, νεολαίας των σοσιαλιστών, όπου χρησιμοποίησε τριών ειδών διαφορετικά όπλα. Και τα τρία αυτά όπλα ήταν στην νόμιμη κατοχή του. Δύο εκθέσεις λοιπόν έχουμε για τις αστυνομικές επιχειρήσεις ε, της αστυνομίας σε ό,τι φορά την 22 Ιουλίου και οι δύο περιλαμβάνουν λοιπόν τέτοια σημαντικά σημεία επίκρισης. Λόγω έλλειψης ακριβώς ε, και απουσίας παρακολούθησης επικίνδυνων ατόμων. Επίσης, ε, περιπτώσεις ψυχασθενών, οι οποίοι διαπράττουν επιθέσεις χωρίς κάποιο πολιτικό κίνητρο, χωρίς κάποιο άλλο σαφές κίνητρο. Ούτε αυτοί λοιπόν εντοπίζονται στο ραντάρ. Και όλη αυτή η δημόσια συζήτηση που λαμβάνει η χώρα στην Νορβηγία έχει αλλάξει είναι πολύ πιο μεγάλη η αποδοχή του γεγονότο ότι η αστυνομία θα πρέπει αναγκαστικά να ξέρει τι συμβαίνει στην Νορβηγία. Γιατί χρειάζονται πολύ απλά πόρου. Υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση λοιπόν για την αστυνομία, υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση για την ανάγκη να παρακολουθεί η αστυνομία τι εξελίξει. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι η Νορβηγία ήταν πολύ αθώα, αν θέλετε, αφελή χώρα. Έχουμε μια κουλτούρα εμπιστοσύνη. Τα τελευταία χρόνια μόλι έχει παρουσιαστεί έντονα αυτή η ανάγκη να μας προστατεύει, για παράδειγμα, η αστυνομία, να προστατεύει η αστυνομία τους πολιτικούς. Okay, right language. Um, thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα αλλάξω ρόλο και ως σκιώδης των φιλελευθερών θα θέσω ορισμένε ερωτήσει, και νομίζω ότι και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι που είναι παρόντες έχουν ζητήσει το λόγο. Υποθέτω και η κυρία Σίπελ θα ήθελε να θέσει ερωτήσεις. Ωραία. Καταρχήν, εγώ να θέσω κάποιες ερωτήσει ως σκιώδης εισηγήτρια εκ μέρους του Άλντεν, των φιλελεύθερων. Έχω τρία σύνολα ερωτήσεων. Καταρχήν, είπατε ότι το σύστημά σας λειτουργεί καλά, θεωρείτε ότι έχετε βαρκή εποπτεία και έτσι όπως το περιγράψατε, ακούγεται πράγματι πολύ αποτελεσματικό. Όμως, ποιες ήταν οι αντιδράσεις σας σε όλες τις αποκαλύψεις μαζικής παρακολούθησης, ιδίως καθώς η χώρα σας βρίσκεται δίπλα στη Σουηδία, που ό,τι φαίνεται είναι ένας από τους κύριους κόμβους σε όλα τα δίκτυα και αν δεν κάνω λάθος, ήδη αυτό εντοπίστηκε από κάποιον ε, που ξεκίνησε την ε, έρευνα. Έτσι λοιπόν όλα αυτά ήταν ορατά σε κάποιο βαθμό. Εσείς έχετε την εντύπωση ότι πρόκειται για κάτι για το οποίο θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί. Δεύτερον, είπατε ότι έχετε εποπτεία επί των εγχώριων, επί των εθνικών υπηρεσιών παρακολούθησης, επί των εθνικών μυστικών υπηρεσιών, αλλά είναι κάπως δύσκολο να μάθετε τι συμβαίνει σε περιπτώσεις της συνεργασίας. Φυσικά αυτά είναι τα κύρια ζητήματα, γιατί ακόμη και αν υπάρχουν μηχανισμοί υποπτήρες που σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ αδύναμοι, τη στιγμή που υπάρχει διασυνοριακή συνεργασία, η συνεργασία αυτή δεν εμπίπτει σε καμία δημοκρατική εποπτεία. Και έχω και κάποιες ερωτήσει για την υπόθεση Breivik. Είπατε ότι τώρα υπάρχει μεγαλύτερη αποδοχή από την πλευρά του κοινού για τη συλλογή των δεδομένων. Αλλά εγώ στον τύπο διάβασα ότι ο Μπρέιβικ ήδη είχε εμφανιστεί στο ραντάρ των αστυνομικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών ασφαλείας. Αυτό είναι ένα μοντέλο που βλέπουμε σε όλες τις μεγάλες επιθέσεις ότι ήδη εκ των προτέρων ήταν γνωστοί οι δράστες στις μυστικές υπηρεσίες. Επομένως, είχαν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και αν ήδη είχε εντοπιστεί ο άνθρωπος αυτός, τότε προφανώς ήδη είχαν τις εξουσίες που χρειάζονταν οι υπηρεσίες ασφαλείας και τα δεδομένα που χρειάζονται. Έτσι λοιπόν, μήπω πρέπει να βελτιώσουμε το την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, αντί να λέμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα βασικά επί αθών πολιτών, γιατί έτσι μεγαλώνει ο σωρός χείρα και δυσκολευόμαστε να εντοπίσουμε τέτοιους ανθρώπους. Και μια τελευταία ερώτηση. Μας ε, έλεγαν πάντοτε ότι η λεγόμενη συμφωνία TFTP ή τα δεδομένα TFTP, η συμφωνία που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι ιδιαίτερα επίμαχη, και που έχει ζητήσει να ανασταλεί το κοινοβούλιο. Μας είπαν ότι ήταν ουσιαστική στην υπόθεση Μπρέιβικ, όχι για την πρόληψη των επιθέσεων, αλλά υποθέτω για την έρευνα και τη δίωξη. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε αν κατά την άποψή σας ε, θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί όπως συμφωνίες αμοιβαίας ε, νομική συνδρομής που υπάρχουν μεταξύ ΗΠΑ και ευρωπαϊκών χωρών, αν κατά την άποψή σας άλλοι μηχανισμοί θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί να ζητηθούν συγκεκριμένες πληροφορίες για μια συγκεκριμένη υπόθεση, αντί να υπάρχει αυτή η χίδη διαβίβαση δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. για την πρώτη ερώτηση. Για το αν μας εξέπληξε ο βαθμός της μαζικής παρακολούθησης. Ναι, βεβαίως. Η κοινή γνώμη στην Ορβηγία αλλά και η πολιτική, δεν γνωρίζουν περισσότερα από ότι ο μέσος αναγνώστης της εφημερίδας. Επομένως, όταν ε, βλέπει κανείς ότι υπάρχουν μυστικοί διευλοί που συνδέουν τον Ορβηγικό κράτος ε, με ε, τους μεγάλες εταιρείες πληροφορικής, και εκεί βλέπουμε να εμπλέκονται εταιρείε πολύ μεγάλες όπως η Apple, η Microsoft, η Google. Και στις Ηνωμένε Πολιτείε δεν θεωρούν ότι πρόκειται για διεθνή παρακολούθηση. Γιατί οι εταιρείε αυτές βρίσκονται σε Αμερικανική δικαιοδοσία και αυτές οι υπηρεσίες ε, όταν τους ζητείτε πρέπει να παραδίδουν τις πληροφορίες. 40.000 ε, τέτοια αιτήματα εστάλησαν στην Google σε σχέση με και ζητούσαν συγγνώμη πληροφορίες σε σχέση με πελάτες της Google. Και νομίζω ότι γενικά αυτό σώκαρε και την κοινή γνώμη και τους πολιτικούς ε, στην Ορβηγία. Στην Ορβηγία έχουμε μια και περίπτωση. Η Σουηδία έχει ψηφίσει ένα νόμο καθιστά νόμιμη την παρακολούθηση όλων των πληροφοριών που κυκλοφορούν μεταξύ Νορβηγίας και Σουηδίας. Ακόμη και τις γραμμές επικοινωνία μεταξύ Νότιας και Βόρειας μπορούν να παρακολουθούν οι μυστικές υπηρεσίες της Σουηδίας γιατί υπάρχουν μέσα από τη Σουηδία. Δηλαδή, οι μυστικές υπηρεσίες της Σουηδίας μπορούν να υποκλέπτουν τηλεφωνήματα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαβιβάζονται από το ένα μέρος της Νορβηγίας στο άλλο. Και προφανώς αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για ένα κυρίαρχο κράτος. Η εθνική κυριαρχία δεν είναι ένα θέμα μόνο φυσικών συνόρων και παρακολούθησης του ποιος ε, περνάει τα σύνορά σου, αλλά έχουμε και κάποια εικονικά σύνορα και σε ένα κυρίαρχο κράτος μόνο η δική του κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε παρακολούθηση των δικών της πολιτών για να δει αν προβαίνουν σε κάποια δραστηριότητα που ενδιαφέρει την αστυνομία. Πρόκειται για μια αρμοδιότητα που έχει αναθέσει στη δική σου αστυνομία. Δεν μπορεί να την αναθέσει σε ένα άλλο έθνο. Ακόμη και αν είναι φιλικό το έθνο αυτό και με τη Σουηδία έχουμε φιλικέ σχέσει, είμαστε εταίροι σε πολλά επίπεδα. Όμως, ε, τελικά, οι νορβηγικές αρχές είναι αυτές που πρέπει να ασχολούνται με τους νορβηγούς πολίτες. Και έχουμε τώρα και μια νέα κυβέρνηση στην Νορβηγία και έχει τεθεί στο πρόγραμμά τους ε, και το θέμα της σουηδικής ε, νομοθεσίας, της λεγόμενη, του λεγόμενου νόμου ΕΦΑ, όπως λέγεται. Αυτή η νομοθεσία δίνει στους ε, Σουηδούς την δυνατότητα να παρακολουθούν τις νορβηγικές τηλεπικοινωνίες. Όταν μιλάμε για διασυνοριακή συνεργασία, πάντοτε τίθενται προβλήματα εκεί, αλλά πρέπει να σεβόμαστε την εξή αρχή. Δεν μπορεί κανείς να παραδώσει σε ξένες μυστικές υπηρεσίες, να δώσει σε ξένες μυστικές υπηρεσίες το δικαίωμα να μπουν στα δικά σου προγράμματα επικοινωνιών και να αντλήσουν από εκεί δεδομένα. Αυτό πρέπει να το κάνουν οι τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες. Ό,τι αφορά τώρα την υπόθεση δεν υπήρχαν ιδιαίτερα προβλήματα στην έρευνα. Ομολόγηση, υπήρχαν και μάρτυρες, υπήρχε ακριβής περιγραφή για τις πράξεις του. Έτσι λοιπόν από τη σκοπιά της έρευνας ε, δεν υπήρχε ιδιαίτερη ανάγκη να προστρέξουμε στις μυστικές υπηρεσίε. Όμως το ερώτημα ήταν ε, αν οι μυστικές υπηρεσίε της αστυνομίας θα έπρεπε να έχουν εντοπίσει και να προλάβουν αυτή την εξέλιξη πριν γίνουν δηλαδή αυτές οι τρομακτικές επιθέσεις. Είναι αλήθεια ότι ο κ. Πλέδικ είχε πυρικό μητρό είχε βέβαια καταδικαστεί για βανδαλισμό, ότι το διάγραψε ένα σύνθημα στον τοίχο, όχι για τρομοκρατία. Έτσι λοιπόν, αυτό ήταν και ένα ακόμη λόγο που δεν είχε εμφανιστεί στα ραντάρ τη αστυνομία. Ήταν ένα μοναχικό λύκο. και πολύ συχνά είναι πολύ δύσκολο να τους εντοπίσεις ε, αυτούς τους ανθρώπους γιατί δεν ανήκουν σε κάποιο κύκλο Τώρα, για το άλλο άτομο που αναφέρατε. Α, συγγνώμη, για το έσελον που αναφέρατε. Έχουμε προχωρήσει πολύ πέρα από το έσελον και έχουμε τώρα την νομοθεσία FRA στη Σουηδία που θέτει πολύ μεγάλο πρόβλημα για μας ό,τι αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Okay, next speaker on... Ωραία. Έχω τέσσερις, ε, ο κυρία Μόρβα, ο κύριο Ζήμπο, ο κύριο Άγκστρομ και ο κύριος Η Κυρία Μόρβα. Ε, ε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω ουγγρικά με την ευκαιρία. Είναι η μητρική μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το φίλο από την Ορβηγία για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Πρώτη ερώτηση. Εάν αυτή η υπόθεση υποκλοπών σόκαρε το κοινό όταν αποκαλύφθηκε, επειδή ήταν πολύ πιο ευρύ από ό,τι κανείς περίμενε και δεν έχει να κάνει πλέον και με την εθνική ασφάλεια, τότε πώς γίνεται εκ μέρους εκείνων που λαμβάνουν τις αποφάσεις να επιδείχθηκε τόσο λίγο ενδιαφέρον για το τι θα μπορούσε να γίνει για κάτι τέτοιο. Από τα 80 μέλη του Κοινοβουλίου, μόνο τέσσερα είμαστε εδώ που δείχνουν ενδιαφέρον και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Για να παραφράσω το ερώτημα, μάλλον είχε δίκιο ο κύριος Σνόουντεν και αυτό που φοβόταν θα πραγματοποιηθεί. Δηλαδή, η αποκάλυψη της αλήθειας μπορεί να μην οδηγήσει πουθενά παρόλο που ρίσκαρε τη ζωή του για να αποκαλύψει την αλήθεια. Η επόμενη ερώτησή μου. Αν οποιοδήποτε κράτος μέλος σαν το δικό σας που επιλαμβάνεται του ελέγχου και της παρακολούθησης ε, των ε, μυστικών υπηρεσιών ε, ή του, των υπηρεσιών του στρατού και της αστυνομίας, αν προσπαθώντας να προστατέψει τα δικαιώματα των πολιτών έναντι τέτοιων παραβιώσεων των δικαιωμάτων, αν Υπάρχει ένα τέτοιο ε, σύστημα ελέγχου λοιπόν. Πώς ε, θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνει θύμα των ε, αντιμαχιών μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και θα ασχοληθεί με την προστασία των πολιτών έναντι της κατάχρησης εξουσίας. Το τρίτο ερώτημά μου όσον αφορά στους ε, ανθρώπους που διαμαρτύρονταν μπροστά από την Αμερικανική Πρεσβεία στο Όσλο. Αυτό λίγο με, έκανε να επιστήσω την προσοχή μου σε αυτό το θέμα. Από ό,τι κατάλαβα από αυτά που είπατε, έπρεπε η Επιτροπή EOS να εξετάσει το θέμα. Αν σας κατάλαβα καλά, ήταν άνθρωποι που διαμαρτύρονταν μπροστά στην Πρεσβεία στο Όσλο. και οι μυστικές υπηρεσίες τους παρακολούθησαν. Ε, και κάποιες από τις διαδικασίες ήταν παράνομες. Πώς φτάσατε σε αυτό το συμπέρασμα, ποιες ήταν αυτές οι παράνομες διαδικασίες και υπήρξε δημόσια καταβρα... κατακραυγή μετά από αυτό, όταν αυτό αποκαλύφθηκε. Επειδή είμαι από μία πρώην κομμουνιστική χώρα, ε, θα θεωρούσαμε ότι σε μια δημοκρατική χώρα της Δύσης αυτό δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβεί, αλλά από ό,τι φαίνεται συμβαίνει. Κύριε Τέτσνερ. Ευχαριστώ. Όσον αφορά στην πρώτη ερώτησή σας, γιατί εκπλήσεστε. δεν υπάρχει μεγάλη πίεση από την κοινή γνώμη να μην υπάρχει παρακολούθηση. Αν η κοινή γνώμη δει ότι κάτι τους πλήττει προσωπικά, τότε μόνο πραγματικά θεωρούν ότι είναι σημαντική η παρακολούθηση και την επιζητούν. Πολλές φορές θα συζητάμε τα θέματα αυτά στην τηλεόραση. Υπάρχουν 5.000 κάμερες στην πόλη του Όσλο. Ξεκίνησε ε, ως ε, ένα αμφίβολο project, αλλά τελικά ο κόσμος είδε ότι μειώθηκε το έγκλημα στους δρόμους και ο καθένας κατάλαβε ότι δεν έχει κάτι να κρύψει. Αυτό προφανώς εξηγεί το γεγονός ότι κανείς πλέον δεν υποστηρίζει δυναμικά και πολιτικά την άποψη να αποσυρθούν αυτές οι κάμερες. Εγώ θεωρώ ότι το θέμα αυτό από πολιτική άποψη δεν έπρεπε να είναι ένα θέμα αντιπαράθεσης. Γι' αυτό έχουμε μία μη πολιτική επιτροπή EOS. Αναφέρονται στους ερετούς πολιτικούς, τα μέλη δηλαδή του Κοινοβουλίου στην Επιτροπή την Κοινοβουλευτική όπου συζητούμε ε, με βάση τη συνένεση. Δεν είναι θέμα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Είμαστε όλοι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι. Η επόμενη ερώτηση είχε να κάνει με την ε, αμερικανική περίπτωση για την παρακολούθηση της περιοχής γύρω από την πρεσβεία της Αμερικής. Αυτό το θέμα δεν έχει τελειώσει. Δεν ξέρω τι θα κάνει η Επιτροπή EOS τελικά. Δεν με τα συμπεράσματα. Από ό,τι φαίνεται η Αμερικανική Πρεσβεία παρακολουθούσε τους δρόμους γύρω από την πρεσβεία. Όχι μόνο όσους ε, κάναν διαμαρτυρία, τους διαδηλωτές έξω από την πρεσβεία. Ευχαριστώ κυρία Ζήπη. Ευχαριστώ. Έχω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Στην αρχή της ε, εισαγωγής σας είπατε ε, γιατί δημιουργήθηκε το 1996 αυτό το ε, Συμβούλιο Ελέγχου και αναφέρατε και κάποια παραδείγματα και κάποια σχετικά, κάποιες σχετικές αφορμές. Ερωτώ λοιπόν, σε ό,τι αφορά την νορβηγική αριστερά αυτή, ήταν δραστηριότητα αυτή της, ε, των μυστικών υπηρεσιών, ήταν δική τους πρωτοβουλία ή υπήρξε πολιτική εντολή άλλων αρχών, της κυβέρνησης για παράδειγμα. Υπήρξε συγκεκριμένη ε, αφορμή για την παρακολούθηση αυτή θεωρήσαμε ότι α, είναι αριστερή αυτή να τους ελέγξουμε για να είμαστε σίγουροι. Και σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις δηλαδή στις σημερινές ε, υπηρεσίες υπάρχουν ε, κάπου περιγραφή των καθηκόντων, των δικαιωμάτων, τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν αυτές οι μυστικές υπηρεσίες. Αν δεν υπάρχει τέτοια περιγραφή, επί ποιας βάσης κάνετε εσείς ελέγχους Πώς αξιολογείτε τα ευρήματά σας, τα πορίσματά σας, αν δεν υπάρχει μια τέτοια βασική περιγραφή των καθηκόντων. Και ύστερα, από το 96 και μετά, οι καταγγελίες των πολιτών έχουν αυξηθεί ή μειωθεί και επίσης το ήτος των καταγγελιών, οι τομεί δηλαδή στους οποίους κινούνται έχουν αλλάξει. Τέλος, με τελευταία ερώτηση πριν από πολλούς μήνες, πριν από χρόνια, κάναμε μία συζήτηση εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων. Και νομίζω ότι ένας συνάδελφος ε, ανέφερε το Minority Report, μία ταινία. Στη συζήτηση λοιπόν αυτή μου θυμίζει όλη η συζήτηση την ταινία αυτή, το Minority Report. Γιατί έχω την εντύπωση ότι οι μυστικές υπηρεσίες κάνουν αυτό που περιγράφεται στην ταινία. Δηλαδή, προσπαθούν να συλλέξουν όσο πιο πολλά δεδομένα γίνεται για το όσο πιο πολλού πολίτε όσο πιο πολλέ οργανώσεις γίνεται και βάσει των δεδομένων αυτών προσπαθούν να κάνουν μια πρόβλεψη για το κατά πόσον θα συμβεί ένα έγκλημα ή όχι. Αν μου πείτε ότι όχι, κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι εμείς πάντα έχουμε ένα συγκεκριμένο ύποπτο, μια συγκεκριμένη ένα συγκεκριμένο λόγο για την παρακολούθηση. Αυτό θα με καθεσύχαζε, αλλά για πείτε μου κατά πόσον παίζει αυτή η μεθοδολογία κάποιο ρόλο στην δουλειά Σα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε να απαντήσει, λέει η πρόεδρο. Σας ευχαριστώ. Το 1996, τι συνέβη. Συνεχίστηκε αυτή η λογική του ψυχρού πολέμου. δεν ήταν τόσο το θέμα το ότι καταδιώξαμε τους, τους κάποιες ομάδε πολύ, ομάδες και πολιτικά αριστερά κόμματα. Υπήρχαν διάφορες δραστηριότητε φυσικά στην, στο αριστερό κόμμα τότε. Αλλά η άποψη που επικρατούσε τότε ήταν η εξή. Αν κάποιος μία ολόκληρα μια ολόκληρη ζωή προσπαθεί να βγάλει την Νορβηγία από το ΝΑΤΟ, κατά πάσα πιθανότητα τα άτομα αυτά θα είχαν και άλλους στόχους πέρα από αυτούς τους πολιτικούς στόχους. Το θέμα λοιπόν ήταν ε, το υπέρ ή κατά του ΝΑΤΟ. Και μιλάμε για οργανώσεις της άκρας αριστεράς. Ακραίες ακραίε σε σχέση με το από παραδοσιακό αριστερό κόμμα του εργατικού. Αποτελούσαν κίνδυνο για την πολιτική ασφαλεία τη Νορβηγία. ήταν πραγματικά υπερβολικέ αυτέ οι δραστηριότητε του. και αυτή ήταν αυτό το πόρισμα τη έκθεση τη Επιτροπή Λάντ όπω ονομάστηκε. Να τονίσω όμω το πλαίσιο αυτό ότι υπάρχουν συγκεκριμένε διαδικασίε. για την παρακολούθηση των πολιτών. αν θέλει κανείς να υποκλέψει τηλεφωνικές συνομιλίες, να παρακολουθήσει τον κόσμο στα σπίτια του, να ανοίξει επιστολές, χρειάζεται δικαστική απόφαση. Και τι κάνει λοιπόν η Επιτροπή, αξιολογεί κατά πόσον η αστυνομία ξεπέρασε ή όχι τα ωριά της. Οι μυστικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες ασφάλειας χρειάζονται δικαστική απόφαση για να εκτελέσουν τις ενεργείες αυτές. για τις καταγγελίες. Όπως σας είπα, περίπου 20 τέτοιες καταγγελίες γίνονται ετησίως. Κάποιες εξ αυτών προέρχονται από άτομα που έχουν ιατρικό ιστορικό και έτσι λόγω του προσωπικού τους υποβάθρου δεν είναι τόσο ουσιώδεις ε, αυτές οι καταγγελίες. Περίπου 15-20 από τις καταγγελίες αυτές, ε, λοιπόν, είναι άτομα που έχουν κάποιο ιατρικό πρόβλημα, που λένε ότι τους παρακολουθούν. Ε, και λίγο πολύ, να σας πούμε την αλήθεια, είναι λίγο παρόμοιο το περιεχόμενο των καταγγελιών αυτών πάντα. Ο αριθμός των καταγγελιών τώρα, ο συνολικός αριθμός, λίγο πολύ είναι σταθερός κάθε χρόνο. Και συμφωνώ μαζί σας ότι μπορεί κανείς ε, τελικά να υπερβάλλει σε ό,τι αφορά την ε, συλλογή των δεδομένων και τελικά βρίσκεται κανείς αντιμέτωπος με ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών που δεν έχει δυνατότητα να το αξιοποιήσει. Ε, ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ. Θα θέσω μια ερώτηση στα σουηδικά. Όπως ε, είπατε, οι νορβηγικές αρχές δεν μπόρεσαν ε, να αποτρέψουν το Πρέδικ ε, από αυτές τις τρομερές επιθέσεις. Είπατε ότι ένας από τους λόγους που λαμβάνει η παρακολούθηση των νορβηγών πολιτών ε, είναι για να σταματήσουν να γίνονται τέτοιες επιθέσεις. Έχουν υπάρξει άλλες περιπτώσεις όπου μπορέσατε να προλάβετε μια τρομοκρατική επίθεση. Ξέρω ότι η Νορβηγία είναι ένα κράτος δικαίου, δεν προβαίνει σε τέτοιες παραδόσεις κτλ. Επομένως, αυτό που θέλω να ρωτήσω, αυτή η παρακολούθηση βοήθησε να βρείτε κάποιον που προετοίμαζε μια τροποκρατική επίθεση και μπόρεσε να δικαστεί στην Ορβηγία. Μια άλλη ερώτηση. Η Σουηδία και η Νορβηγία ανταλλάσσουν ε, πολλές πληροφορίες και στρατιωτικού και μη στρατιωτικού χαρακτήρα και όπως είπατε η Σουηδία έχει μια νομοθεσία ε, που της δίνει το δικαίωμα να παρακολουθεί τους νορβηγούς πολιτούς όσο θέλει, ανεξαρτήτως με το αν αυτό ή όχι. Επομένως, ο νόμος αυτός της Σουηδίας σας έχει βοηθήσει να καταδικάσετε τρομοκράτες ή να προλάβετε κάποιες τρομοκρατικές επιθέσεις. Απάντηση για το πρώτο σχόλιο σας. Ένας από τους λόγους για τον οποίο δεν παρακολουθούμε τις δραστηριότητες των ιδιωτών είναι ότι δεν μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε τις δράσεις του ατόμου αυτού, όμως ε, αυτό που μας κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν ε, οι ποσότητες που είχε παραγγείλει και τα κύρια συστατικά της βόμβας είχαν καταγραφεί από τις μυστικές υπηρεσίες, όμως ήταν λογικό να έχει παραγγείλει τέτοια υλικά κάποιος που σχολόταν, που δραστηριοποιούταν ε, στο επάγγελμα αυτό και σε ό,τι αφορά τώρα τη σουδική νομοθεσία δεν μας βοήθησε γιατί κανένας και στην Νορβηγία δεν θα μπορούσε να έχει προλάβει την επίθεση αυτό. Έτσι λοιπόν μπορώ να απαντήσω αρνητικά. Δεν ξέρω αν η δεύτερη ερώτησή σας απαντήθηκε πλήρως. Αν ε, αποτράπηκαν κάποιες επιθέσεις. Νομίζω ναι, απαντήθηκε ότι ε, μυστικές ε, υπηρεσίες ε, της ε, Νορβηγίας κατέληξαν στο μηδέν και το ίδιο ισχύει και για τις Σουηδικές υπηρεσίες. Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Ο κύριος Έντσιου, ο οποίος δεν είναι εδώ από ό,τι φαίνεται, μάλιστα. Και εδώ κλείνουμε τη συζήτηση αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ διαφωτιστική η παρέμβασή σας. Σας ευχαριστούμε που παρευρεθήκατε εδώ. Έτσι λοιπόν περνάμε τώρα στο δεύτερο τμήμα της συζήτησης, στην παρουσίαση του πρώτου εγγράφου εργασία ε, για τις δραστηριότητες παρακολούθησης των ΗΠΑ ε, σε σχέση με τα δεδομένα, τα ευρωπαϊκά δεδομένα και τις ε, πιθανές νομικές επιπτώσεις στις διεθνωτικές συμφωνίες και τη συνεργασία. Ο κύριος Μουρές δεν είναι εδώ, έτσι λοιπόν θα ζητήσω από τον κύριο Βόξ να παρουσιάσει το έγγραφο και στρέφομαι και προς τη γραμματεία. Δεν υπάρχει έγγραφο στο φάκελο. Προφορική θα είναι η παρουσίαση. Θέλετε να πείτε κάτι. Ναι, σας παρακαλώ, κάτι διαδικαστικό. Γιατί ο κύριος Μωράες ε, δεν είναι εδώ και είναι εισηγητής. Εγώ νομίζω ότι είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει εδώ. Δηλαδή δεν είναι εδώ συγητέ. Ε, δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτησή σα, λέει πρόεδρο. Ε, δεν γνωρίζω εγώ τι κινήσει του κυρίου Μωράε. Είμαι σίγουρη ότι έχει πολύ καλού λόγου που δεν παρευρίσκεται εδώ, όμω δεν μπορώ να σα εξηγήσω. Νομίζω ότι εσεί πρέπει προσωπικά να του θέσετε αυτή την ερώτηση. Δεν είναι προσωπικό το θέμα αυτό, είναι πολιτικό το θέμα, λέει κυρία Μορβάη. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ρωτήσω εγώ γιατί οποιοδήποτε δεν είναι παρόν εδώ. Λυπάμαι. Κύριε Φώση, το λόγο. So, vielen Dank. Ευχαριστώ. Αυτό το πρώτο έγγραφο εργασίας ασχολείται με την παρακολούθηση σχετικά φυσικά με τα δεδομένα, αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις, ειδικότερα τις ε, νομικές επιπτώσεις ε, των υφιστάμενων ε, διατλαντικών συμφωνιών και της συνεργασίας. Πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού, εδώ στην Επιτροπή ε, μάθαμε για όλο αυτό το θέμα του NSA και ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια είδαμε πως ε, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία διαμορφώνονται οι διατλαντικές ε, σχέσεις. Αυτό συνοψίζεται σε αυτό το έγγραφο δεν μιλάμε μόνο για το νομικό πλαίσιο της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν διαφωτίζεται μόνο αυτό, αλλά ε, όλες οι συμφωνίες μεταξύ ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, η ε, CFDP, η ΚΕΠΑ κτλ. Η πρώτη συμφωνία είναι μια οικονομική συμφωνία η οποία έχει ξεκινήσει από την πλευρά των Αμερικανών από το Υπουργείο Εμπορίου και Μεταφορών και, από έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ουσία επιτρέπει να μεταφέρονται νόμιμα δεδομένα στις Ηνωμένε Πολιτείες και αυτή τη στιγμή να υπάρχει αυτή η δυνατότητα και ειδικότερα ε, να μεταφέρονται δεδομένα προσωπικά ανθρώπων σε τρίτες χώρες αν δεν υπάρχει παρόμοιο επίπεδο ασφαλείας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η συμφωνία για το Safe Harbor, το ασφαλές καταφύγιο, ε, ταυτόχρονα διασφαλίζει ότι και οι εταιρείε μπορούν να μπουν σε αυτήν την συμφωνία όταν δεσμευθούν να ε, τηρούν τις αρχές αυτής της συμφωνίας και συγκεκριμένα την προστασία των προσωπικών δεδομένων ε, Ευρωπαίων πολιτών ε, που διασφαλίζεται στις ΗΠΑ και σε τρίτες ε, ε, χώρες. Αυτή η συμφωνία, η Safe Harbor, όλο και περισσότερες κριτικές δέχεται και αυτές οι επικρίσεις έχουν να κάνουν με την εντατικοποίηση της ανάλυσης των δεδομένων, η οποία γίνεται όλο και μεγαλύτερη και όλοι ζητούν να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο έτσι ώστε να αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό. Η ίδια η συνθήκη ε, σε περίπτωση παραβίωσης της ε, ρυθμίζει στο άρθρο 3 ότι θα πρέπει να υπάρχει απόφαση για κατάργησή της ε, από τους συμβαλόμενους και ως αντίδραση στο ε, σκάνδαλο για τις παρακολουθήσεις ε, φέτος το καλοκαίρι η Κομισιόν ξεκίνησε μια αξιολόγηση και την, τελευταία, την περασμένη εβδομάδα μας ε, παρουσίασε και χαίρομαι που συνέβη αυτό μέσα από την ανακοίνωση της Κομισιόν και τις συστάσεις για την βελτίωση της λειτουργικότητας αυτής της συμφωνίας. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αυτή η προσέγγιση που προτείνει η Κομισιόν δεν είναι μια επαρκής λύση γιατί θεωρώ και αισθάνομαι και το είδαμε και για τις παρακολουθήσεις από πολλές πλευρές συμφώνησαν όλοι ότι αυτή η safe harbor, η συμφωνία safe harbor δεν είναι πλέον safe, δεν είναι πλέον ασφαλής. η προστασία των δεδομένων και η αποκάλυψη δεδομένων που γίνεται αυτή τη στιγμή ε, μπορεί να φτάνει στα όρια του παρανόμου από την πλευρά της NSA και από άλλα μέρη, ας πούμε τις εταιρείες ε, που ασχολούνται με αυτά τα δεδομένα και τα συλλέγουν. Με όλο και πιο εντατικό τρόπο αναλύουν τα δεδομένα έτσι λοιπόν μακροπρόθεσμα τα δεδομένα των πολιτών μας θα πρέπει να προστατευτούν καλύτερα. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να έρθει η συμφωνία αυτή, να την θέσουμε σε νέα βάση. Γιατί ε, η συμφωνία αυτή δεν έχει μόνο πολιτικές, αλλά έχει και οικονομικές επιπτώσεις, ειδικότερα για τους οικονομικούς εταίρους, ε, είπα Ευρωπαϊκή Ένωση. μεσοπρόθεσμα θα πρέπει θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι θα πληγούν οι εταιρείες ε, του διαδικτύου και ότι ειδικότερα οι, πολίτε οι πολίτες μας θα πρέπει να λαμβάνονται πιο σοβαρά υπόψη και να προστατεύονται καλύτερα σε επίπεδο προσωπικών δεδομένων, μέχρι δηλαδή να βρούμε ε, μια νέα μορφή για τη συμφωνία και να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη στη σχέση μεταξύ ΕΕ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ. Τώρα για την ε, συμφωνία TFTP. Είναι πολύ σημαντική για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η συμφωνία έχει να κάνει με το πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και είναι ένα πολύ σημαντικό ε, εργαλείο για την πάταξη της τρομοκρατίας και των μεγάλων εγκλημάτων, των σοβαρών εγκλημάτων. Για παράδειγμα, θα βοηθούσε και σε μια περίπτωση σαν αυτή του Μπρέιβικ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Θεωρεί ότι πρέπει σε, αυτό το, σε αυτή τη συμφωνία πρέπει να υπάρχει χρυσή τομή μεταξύ της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ε, θέλουμε όσο, και, όσο περισσότερο γίνεται να προστατεύεται η προσωπική σφαίρα των ανθρώπων. Με αυτή την ε, άποψη συνταχθήκαμε και ήμασταν υπέρ αυτής της συμφωνίας, γιατί θεωρήσαμε ότι θα παρακολουθεί τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια στανταρά ασφαλείας που θα σχετίζονται με αυτήν τη συμφωνία. Σύμφωνα με το άρθρο 121 είναι δυνατή η καταγγελία αυτής της συμφωνίας. Στις 23 Οκτωβρίου έγινε ένα αίτημα από την πλευρά του ΕΛΚ και στην Κομισιόν να καταγγελθεί αυτή η συμφωνία λόγω της παραβίασής της, ε, σύμφωνα με το άρθρο 121 δηλαδή, ε, να ληφθούν μέτρα. Η Επίτροπος Μάλστρομ την περασμένη εβδομάδα ήρθε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και μας ε, ενημέρωσε και είπε ότι σε συνεργασία με τη ΣΥΠΑ είδε ότι ε, η Κομισιόν δεν έχει στοιχεία για παραβίαση της συμφωνίας από την NSA. Εμείς στην ακρόαση με την Ευρωπόλ και με την SWIFT, την εταιρεία SWIFT, αυτή μας είπε ότι δεν έχει στοιχεία, όμως θεωρώ ότι οι ε, οικονομικές ε, επιπτώσεις της τρομοκρατικής επίθεση της 11 Σεπτεμβρίου ήταν μια εξαιρετική σημασίας και οδήγησαν σε ε, αυτή τη στρατηγική για την παρακολούθηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Όμως η Κομισιόν δεν ανταποκρίθηκε τα όσα είχαμε πει τότε για ένα νομοθετικό πλαίσιο και ένα τεχνικό πλαίσιο για την εξέβρεση και αξιολόγηση των πληροφοριών. Με το πρόγραμμα αυτό, το TFTP, στην ουσία προσπαθούμε να εξισορροπήσουμε την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων και να το κάνουμε αυτό σε συνεργασία με τη ΣΥΠΑ. Άρα, αν αρθεί αυτό το πρόγραμμα, δεν θα εξυπηρετηθεί αυτός ο στόχος. Από τη μία, τίθεται υποαμφιβόλο η ασφάλεια των πολιτών μας και από την άλλη αναρωτιόμαστε πώς γενικά θα πρέπει μέσα σε αυτά τα πλαίσια να έχουμε συμφωνίες με ε, τις Ηνωμένες Πολιτείες όταν δεν έχει γίνει αυτό σε αυτή την περίπτωση. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε μια ισορροπημένη σχέση με τον αντισυμβαλόμενο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι ανακαλούμε τη συμφωνία όχι γιατί δεν μας αρέσει ή γιατί το κάνουμε για ε, εκβιασμό. Η τρίτη συμφωνία με την οποία θα ασχοληθώ είναι αυτή για τα δεδομένα των πτήσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΕΠΑ και σε ό,τι αφορά τη μεταφορά τέτοιων ε, προσωπικών δεδομένων των επιβατών ε, που συλλέγουν οι εταιρείε από τους επιβάτες κατά την κράτηση και χρησιμοποιούνται από ένα ε, πρόγραμμα υπολογιστή για τις κατήσεις εδώ η σύμβαση στο άρθρο 24 προβλέπει σε περίπτωση παραβίασης ε, των ε, συνθήκων μία ρήτρα αποχώρησης, μία ρήτρα κατάρχησης, αλλά δεν υπάρχει άλλη υπόδειξη σε περίπτωση κατάχρησης των δεδομένων από τις μυστικές υπηρεσίες. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια εκθέση αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και πάλι αναφέρεται με σαφήνεια ότι σε 23 περιπτώσεις PNR, δεδομένων PNR, 23 δηλαδή υποθέσεις που είχαν δοθεί σε στοιχεία δεδομένα PNR ε, στην NSA, υπήρχαν αμφιβολίες και σε ό,τι αφορά, μάλλον και εξυπηρετούσαν την ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άρα υπήρχε νομική βάση και συνάδουν με τη συμφωνία αυτή. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θα ήθελα να αναφέρω τα στοιχεία αυτό και θα ήθελα να πω σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προσωπικά αυτά δεδομένα, τους φακέλους των επιβατών, θα πρέπει να κοιτάξουμε να καταλήξουμε κι εμείς προς μία ενιαία τέτοια συμφωνία για να μην έχουμε 28 διαφορετικά συστήματα PNR. Συνοψίζοντας, άρα, να πω ότι η αντιμετώπιση των προσωπικών δεδομένων στην ΕΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαφορετικός ο τρόπος αντιμετώπισης των στοιχείων αυτών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται μια θεματοποίηση οριζόντιος και θεωρείται θεμελιώδες δικαίωμα του ατόμου, ενώ στη ΣΥΠΑ έχει να κάνει πιο πολύ με την προστασία του καταναλωτή. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο προσπαθούμε να δώσουμε δικλείδες ασφαλείας και νομικές ε, διασφαλίσεις, ενώ από πλευράς της Αμερικής ε, φαίνεται ότι επικρατούν πιο πολύ οι ανησυχίες για την ασφάλεια. Για το ίδιο το σκάνδαλο υποκλοπών, ασφαλώς και έχει επιπτώσεις στην ιδιωτική σφαίρα των ε, Ευρωπαίων πολιτών, αλλά ουσιαστικά πρέπει να πούμε ότι επιβαρύνει και τις διατλαντικές σχέσεις, οι οποίες σήμερα βρίσκονται σε φάση διαπραγμάτευσης νέων συμφωνιών, όπως το Safe Μπορεί να συνεχίσει τη διαπραγμάτευσή τους, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και μια σωστή αντίδραση. Τώρα, η καταγγελία από πλευράς μας του Safe Harbor νομίζω ότι μπορεί να ενίσχυε τη θέση μας. Δεν ξέρω τώρα για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης τι θα μπορούσε να γίνει να πω ότι σε ό,τι αφορά την ε, συμφωνία πλαίσιο θα πρέπει να φροντίσουμε να την ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατό ένα θέμα το οποίο θα το φροντίσει ο Φίλιπ Λάμπριχτ. Θεωρώ ότι μπορούμε να συμβάλλουμε τα μάλα σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων στο αστυνομικό και δικαστικό πλαίσιο, αλλά και σε ό,τι αφορά το καλύτερο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και να δώσουμε έτσι στους Ευρωπαίους πολίτες τη δυνατότητα να μπορούν να κινηθούν δικαστικά και στη ΣΥΠΑ σε ό,τι αφορά περιπτώσεις κατάχρησης των προσωπικών δεδομένων. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Έχω τρεις, ε, τρία άτομα που ζητούν το λόγο. Zipper, Μόρβαϊ, Έγκστρον. Κανείς άλλος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται έτσι ο κατάλογος των ομιλητών και εγώ θα είμαι η τελευταία ως σκιώδες, η κυρία Zipper. Zipper. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να αναφέρω τα πράγματα στη σειρά που τα ανάφερε και ο συνάδελφος Φως, έτσι όπως μας τα παρουσίασε. Θα ήθελα καταρχάς να κάνω μια πολύ μικρή ερώτηση για τη Συμφωνία Safe Harbor. Η σύσταση είναι να σταματήσει η τρέχουσα διαπραγμάτευση της συμφωνίας να γίνει μια νέου, εκ νέου διαπραγμάτευση. Γιατί να γίνει εκ νέου διαπραγμάτευση, γιατί ευκρινίστε μας κοιτώντας το μέλλον. Ψηφίσαμε το πακέτο για την προστασία των δεδομένων, επιτέλους Μάλλον αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά εάν τα καταφέρουμε και το ολοκληρώσουμε αυτό, γιατί να το χρησιμοποιήσουμε, γιατί να μας ε, χρησιμεύσει η Συμφωνία Safe Harbor σε κάτι. Αυτό είναι σημαντικό για τι νομικέ επιπτώσει. Τώρα για τι νομικέ επιπτώσει τη υπόθεση υπόθεσης NSA. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να τι δούμε ξεχωριστά από το πολιτικό πλαίσιο και είμαι κάπω ενοχλημένη. Σα το ομολογώ. Όταν αναφέρεται ότι η κατάργηση της συμφωνίας TFTP πει δεν θα πρέπει να αποτελεί αντίμετρο, αν θέλετε, εκδίκηση προς τις ΗΠΑ. Κοιτάξτε, εδώ από όσο γνωρίζω πρόκειται για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Απέτηση να ανασταλεί η διαπραγμάτευση της συμφωνίας. Για να σταλεί η συμφωνία. Τώρα να αναφέρουμε και να κρίνουμε την απόφαση του Κοινοβουλίου, τι να σας πω, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι σωστό, ιδιαίτερως στο παρόν ε, συγκείμενο και θεωρώ ότι ως κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να ε, αυτοκατηγορούμαστε. Θα πρέπει να, ε, να υποστηρίζουμε τις αποφάσεις του κοινοβουλίου τώρα. Θα ήθελα να πω ότι από τότε που υπάρχει αυτή η συμφωνία πάντα γίνεται η συζήτηση για το κατά πόσο η συμφωνία η FTP έχει πραγματικά αντίκτυπο στην πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων σε ό,τι αφορά και τις άλλες πτυχές ε, του TFTP, του συστήματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Δεν θα ήθελα να επίσης σε λεπτομέρειες στην παρούσα φάση. Αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάνει λεπτομερή έκθεση ούτε παρακολούθηση για το κατά πόσον το SWIFT ε, πέρα από τη συμφωνία κάλεσε, παραβίασε τη συμφωνία. Η εταιρεία η οποία συλλέγει τα στοιχεία TFTP λέει ότι δεν διαπιστώθηκε επίθεση στον εξυπηρετητή της. Αυτό τι σημαίνει, δεν σημαίνει και τίποτα. Μπορεί να γίνουν και επιθέσεις μεταξύ δύο σερβερ, δύο εξυπηρετητών, η Europol, η υπηρεσία κυβερνοεγκλήματος, αναρωτιέμαι γιατί δεν ζήτησαν πιο πολλές διευκρινήσεις, πιο πολλές πληροφορίες. Απλά έχουμε εμπιστοσύνη ότι α, όλα θα πάνε καλά. Υπάρχουν όμως ε, νομικές επιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα των επιβατών, το φάκελο επιβατών, είπατε ότι θέλουμε να αποφύγουμε την κατάσταση στην οποία θα έχουμε 28 διαφορετικές συμφωνίες. Εγώ καταρχάς δεν πιστεύω να, να συμμετέχουν ενεργά όλα τα κράτη-μέλη σε μια διαδικασία διαμόρφωσης μιας τέτοιας συμφωνίας. Και αν το κάνουν αυτό, από πού το χρηματοδοτούν. Την ε, προηγούμενη εβδομάδα μας είπε η κυρία Μάλμστρεμ ότι δεν θέλουν... Δεν θέλουμε να αναπτύξουμε τα δεδομένα TFTP εδώ στην Ευρώπη, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό αυτό το project. Αυτό λοιπόν είναι που είχαμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το σύστημα PNR, από πού το χρηματοδοτούμε, που θεωρώ ότι δεν έχει και οποιοδήποτε όφελος. Και επίσης να επισημάνω ότι το θέμα του ωφέλους, της χρήσης των δεδομένων για την καταπολεμώση της τρομοκρατίας είναι άκρος αμφιλεγόμενη. Να μην πιστεύουμε και τον τύπο. Η δυνατότητα χρήσης των δεδομένων αυτών περιγράφεται και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγχουμε κατά πόσον υπάρχει νομική παραβίαση της συμφωνίας, κατά δεύτερον και επίσης σημαντικό, κατά πόσον θα πρέπει να αμφισβητήσουμε το σύνολο της συμφωνίας. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση που πραγματικά θα πρέπει εντελεχέστατα να συζητήσουμε τα δύο αυτά θέματα. Ευχαριστώ πολύ, Λίπρατος, κύριε Μορβάη. Ε, Ευχαριστώ. Αν κατάλαβα καλά, τώρα εξετάζουμε ένα σχέδιο έκθεσης ε, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ χωρίς την παρουσία του εισηγητή και ακούσαμε την παρουσίαση του σκιώδους εισηγητή. Ο τίτλος ε, αναφέρεται στις δραστηριότητες παρακολούθησης των ΗΠΑ σε σχέση με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι πιθανές νομικέ επιπτώσει για τις διατλαντικέ συμφωνίες και τη συνεργασία. Ο σκιώδη εισηγητή, καθώς ε, ο εισηγητή αποσιάζει και δεν μπορούμε να μάθουμε την άποψή του, είπε τα εξή. Αφενός, ότι δεν θεωρεί σόφρον σύμφωνα με πληροφορίες της Κομισιόν, μάλλον θεωρεί ότι έχει υπάρξει σοβαρή υπεραβίαση από τις Ηνωμένες σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Δηλαδή, από τότε που ασχολείται η Επιτροπή μας με το θέμα αυτό, δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό που Σνόντεν, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών έχουν πει. Ποια διαδικασία έχουμε ακολουθήσει η Κομισιόν, έχει ανακρίνει το Σνόντεν και εμείς γιατί δεν έχουμε ανακρίνει το Σνόντεν αν και έχω καταθέσει σχετική πρόταση. Θα θέλαμε να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δηλαδή, τι έχει επιβεβαιωθεί, ποια είναι τα γεγονότα και ποιες είναι οι νομικές επιπτώσεις. Ποιο είναι το συμπέρασμα της Κομισιόν και ποια είναι η πρότασή της. Αν κατάλαβα καλά, τίποτα δεν έχει υποθεί ως προς αυτή την κατεύθυνση. Για το αν μπορούμε να προβούμε σε ένα αναστολή των διατλαντικών συμφωνιών. αλλά έχω την εντύπωση ότι όταν εξετάζουν τέτοια ζητήματα, ζητήματα 4-5 από εμά είναι μόνο παρόντε και τελικά δεν θα υπάρχουν επιπτώσει. Λέμε ότι η ένα τμήμα ε, του δυτικού κόσμου, το 1% ε, παρακολουθεί το υπόλοιπο 99% και δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή και οι δυτικές χώρες και οι δικές μας χώρες μπορούν να κάνουν το ίδιο και δεν υπάρχει αντίρρηση γιατί όλοι το θεωρούν φυσικό. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω το Σκιώδη, έχω δίκιο. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου πόσο μακριά έχει φτάσει αυτή η Επιτροπή και ποια θα είναι το περιεχόμενο της έκθεσης που θα δημοσιευτεί τον Ιανουάριο. Πρόεδρος, πριν να δώσω το λόγο στον κύριο Έξτρομ, να σας ενημερώσω κύριο Μορβάη, Η διευθέτηση για την Επιτροπή αυτή είναι εξή. Ο εισηγητή ε, και ο ε, θα καταρτήσουν από κοινού μια έκθεση. Ο κύριο Βό είναι ο σκιώδη ε, εισηγητή εκ μέρου του ΕΛΚ για αυτήν την επιτροπή, αλλά επίσης ε, συνυπογράφει το εγγραφό αυτό. Έτσι λοιπόν ε, θα συγγράψει και αυτός τμήμα της τελικής έκθεσης. Επομένως δεν ε, ακούσατε ένα σχόλιο από οποιοδήποτε σκιώδη συγητή, αλλά από ένα σκιώδη συγητή που θα συντάξει και αυτός το έγγραφο. Κύριο Σέξτρομ, ευχαριστώ. Δυστυχώς ε, δεν ε, έχω στη διάθεσή μου. Δεν ε, μπορείτε γιατί δεν έχει διατεθεί ακόμα και θα είναι στη διάθεσή σας πριν από την Πέμπτη. Τη συνεδρίαση μας της Πέμπτη. Σίγουρα εσύ θα το έχει διαβάσει πάντως. Ναι, δυστυχώς το πρόβλημα είναι ότι δεν φαίνεται να μου στέλνουν αντίγραφα όλων όσων βρίσκουν. Ιδιαίτερα προβληματικό αυτό, αλλά δυστυχώς έτσι λειτουργεί η Λοιπόν, όταν θα έχουμε στη διάθεσή μας το έγγραφο, ελπίζω ότι θα ασκεί μεγαλύτερη κριτική από ό,τι η Κομισιόν, γιατί ναι, κατανοώ ότι η κυρία Μάστρον συνομίλησε με τους Αμερικανούς και είπαν Αμερικανοί, όχι, όχι, δεν παραβιάζουμε καμία νομοθεσία. Και ήρθε η κυρία Μάστρομ, μα είπε, όλα είναι πολύ καλά, δεν έχουν παραβιάσει καμία νομοθεσία. Εγώ νομίζω ότι παρουσιάζεται κάπως αφελής η Κομισιόν εδώ και θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι όταν ρωτάμε τις μυστικές υπηρεσίες για τις δραστηριότητε τους μπορεί και να λένε και ψέματα. Τέλος πάντων αυτή είναι η στάση της Κομισιόν μέχρι τώρα. Και θα ήθελα να έρθω σε ένα παρόμοιο ζήτημα με την ερώτησή μου. Εδώ ακούσαμε από κάποιο προσκεκλημένο μας πόσο αποτελεσματική ήταν η παρακολούθηση της NSA και από ό,τι κατάλαβα υπήρχαν μηδενικές ε, περιπτώσεις ε, όπου τελικά η NSA μπόρεσε να σταματήσει μια τρομοκρατική επίθεση υπόθηκε ότι ήταν, ε, υπήρχε μόνο μία υπόθεση όπου οδήγησε η χρήση αυτών των μαζικών δεδομένων σε καταδίκη στο δικαστήριο, όμως ε, δεν αφορούσε τρομοκρατικά εγκλήματα, αλλά κάποιες οικονομικής φύσεως αδικήματα. Έτσι, λοιπόν, ε, με αυτό το φόντο, η TFT φαίνεται να έχει επιλύσει μηδενικές ε, συνωμοσίες τρομοκρατίας παγκοσμίως. Ακούσαμε και από τη Σουηδία, ακούσαμε και από τα μέλη του ακούσαμε και ότι δεν έγινε τίποτα Στι Ηνωμένε Πολιτείε, το ίδιο θα γίνει και με το PNR, με του καταλόγους επιβατών. Και φαίνεται ότι τελικά όλα αυτά δεν παρέχουν καμία ασφάλεια. Έτσι λοιπόν, μήπω έπρεπε να σκεφτούμε να τα αναστείλουμε εντελώ, να στείλουμε εντελώ όλε αυτέ τι συμφωνίε. Ε, γιατί δεν μπαίνουμε και σε κανένα ιδιαίτερο κίνδυνο να το πράξουμε αυτό, τουλάχιστον εγώ αυτό πιστεύω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και εγώ τώρα με το ρόλο της σκιώδης εισηγήτριας θα πω τα εξής. Δεν θα αναφερθώ στο Safe Harbor, στην περιοχή ασφάλειας, ε, γιατί συμφωνώ με τις απόψεις που ακούστηκαν από τον εισηγητή και την κυρία Σίπελ και άλλους. Σε ό,τι αφορά τώρα το PNR, εγώ ως εισηγήτρια καταψήφισα τη συμφωνία. Δεν έχω αλλάξει γνώμη, το αντίθετο μάλιστα. Νομίζω ότι θα πρέπει και αυτή να ανασταλεί και θα πρέπει να εξετάσουμε και τις άλλες συμφωνίες PNR επίσης. Και παρεπιπτόντω να σα πω ότι δεν νομίζω ότι αυτή η έκθεση έχει καμία σχέση με τα πινάρι τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και δεν μου έδωσε η πρόταση ότι υπάρχει ανάγκη εναρμόνιση μεταξύ 28 εθνικών συστημάτων, γιατί ακόμη δεν υπάρχουν. Και στι χώρε όπου δημιουργούνται, όπω τη δική μου, χωρί νομική βάση, η δημιουργία τέτοιου συστήματο βασίζεται ε, υποστηρίζεται συγγνώμη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ ότι αυτό είναι τρομερικοινικό όμως ε, δεν θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα του Επινάρτη της Ευρωπαϊκής γιατί ότι FTP ε, δεν νομίζω ότι καλούμε για αναστολή ως εκδίκηση, αλλά επειδή πιστεύουμε ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν κρατήσει το λόγο τους, γιατί παραβίασαν τη συμφωνία και επειδή η Κομισιόν ε, είτε δεν είναι πρόθυμη είτε αδυνατή να προβεί σε μια πραγματική έρευνα και να μας παρουσιάσει μια αιτιολογία που να στέκει γιατί δεν προβαίνει στην αναστολή της συμφωνίας. Τέταρτο σημείο, γιατί επικεντρωθήκατε σε αυτές τις τρεις συμφωνίες μόνο γιατί δεν έχετε κεντρωθεί και σε άλλες συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός από το τομέα της ασφάλειας και της επιβολής του νόμου, διμερείς συμφωνίες λόγου χάρη μεταξύ κρατών μελών και Ηνωμένων Πολιτείων, για τη ΦΑΤΚΑ, νομοθεσία για την ε, φορολογική συμμόρφωση και εκεί συλλέγονται πολύ μεγάλοι όγκοι δεδομένων ε, και γιατί δεν ασχοληθήκατε ε, με άλλες συμφωνίες με, όπως με χώρες όπως η Ρωσία υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Europol και Ρωσίας από ό,τι έχω καταλάβει δεν έχει μπει ακόμη σε ισχύ αλλά πρόκειται να γίνει πολύ σύντομα Υπάρχουν και άλλες συμφωνίες με άλλες χώρες πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες που ίσως θα θέλαμε να εξετάσουμε. Κατόπιν, δύο τελικά σημεία. Εδώ πρέπει να προβούμε στην εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων για το μέλλον, κάποια διδάγματα. Καταρχήν, θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη σύναψη διεθνών συμφωνιών και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το δίδαγμα της TFTP. Δηλαδή, όταν έχουμε υπογράψει μια τέτοια συμφωνία, είμαστε εκτός του παιχνιδιού. Αφού το έχουμε κάνει αυτό, είμαστε εκτό του παιχνιδιού. Και εγώ, ω μέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν δίνω λευκέ επιταγέ. Αν δίνουμε την συγκατάθεσή μα σε μια συμφωνία, η ευθύνη μα δεν τελειώνει εκεί. Δεν ε, είμαστε εδώ ε, ένα ρομπότ, μια μηχανή που βάζει σφραγίδες. Πρέπει να δούμε ποιο είναι ο ρόλο Μα Μας ε, έχει δώσει αρμοδιότητε συγκεκριμένε στη συνθήκη για να εγκρίνουμε την σύναψη διεθνών συμφωνιών. Αλλά τώρα, αφού το πράξαμε αυτό, βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι και τόσο πρόθυμη να υπογράψω οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία, οποιοδήποτε είδου. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Και μπορεί να θυμάστε, νομίζω ότι συζητούσαμε την Αμερικανική Συμφωνία PNR, ζητήσαμε τότε από την Κομισιό να δεσμευτεί δημοσίω να παρουσιάσει μια πρόταση για την αναστολή τη λήξη μια διεθνού συμφωνία αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε από την Κομισιόν να το πράξει. Το κάναμε τώρα λοιπόν αυτό και βλέπουμε ότι η Κομισιόν δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί, κοιτάξτε, είμαστε μόνο οι εκλεγμένοι πρόσωποι των 550 εκατομμυρίων πολιτών. Ποιοι είμαστε εμεί να ζητήσουμε τέτοια αναστολή. Επομένω, αυτό οπωσδήποτε πρέπει να αποσαφινιστεί. Και το τελευταίο σχολείο μου. αν επιτρέψουμε τη μαζική συλλογή προσωπικών δεδομένων ή αν υπογράψουμε τέτοια συμφωνίες για τη μαζική παρακολούθηση, τότε η άλλη όψη του είναι η διαφάνεια. Γιατί για μένα η ουσία της δημοκρατίας ε, είναι να υπάρχει ισορροπία, να υπάρχει έλεγχος. Αν ε, δώσουμε κάποιες αρμοδιότητες, κάποιες εξουσίες στις δημόσιες αρχές, πρέπει να δώσουμε και εξουσίες στους πολίτες για να περασπιστούν τον εαυτό τους όταν υπάρχουν λάθη, καταχρήσεις, κάποια αυθαίρετη χρήση της εξουσίας. Και εδώ βλέπετε ότι η νομοθεσία μας δεν επαρκεί Είχαμε ένα κανονισμό σχετικά με τη διαφάνεια, αλλά από ό,τι φαίνεται στην πράξη είναι άχρηστη αυτή η νομοθεσία, γιατί κάθε φορά που υπάρχει οποιοδήποτε αντίκτυπο στις διεθνεί σχέσεις με του φίλου μας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οποιοδήποτε έγγραφο που έχει να κάνει με αυτές τις διεθνεί σχέσεις, σχεδόν αυτόματα χαρακτηρίζεται απόρριτο και εμπιστευτικό. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε το θέμα τη διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το επίπεδο τη διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι απαράδεκτο. Όμω δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε του Αμερικανού για αυτό. Του εαυτού μα πρέπει να κατηγορήσουμε γιατί κάθε φορά δεχτήκαμε τη ρήτρα για εξαιρέσει ε, στον κανονισμό διαφάνεια. Και αυτό βασικά σημαίνει ότι ο κανονισμό περί διαφάνειας είναι καινογράμμα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά, γιατί τώρα εξετάζουμε την αναθεώρηση του κανονισμού διαφάνειας και άκουσα ότι ορισμένε ομάδες εδώ στο Κοινοβούλιο ε, είπαν ότι πρέπει να ολοκληρωθεί όλη αυτή η δικασία πριν το τέλος της θητείας επειδή έχουν τελματώσει οι διαπραγματεύσει. Έτσι λοιπόν ας δεχτούμε χαμηλότερα πρότυπα για τη διαφάνεια, ας υποχωρήσουμε προς το Συμβούλιο και ξεμπερδεύουμε. Εγώ νομίζω όμως ότι είναι πολύ επικίνδυνη η πρόταση αυτή και πρέπει να αντιμετωπιστεί και στο πλαίσιο του κειμένου σας. Αν δεν υπάρχουν άλλα επίγοντα θέματα, να δώσω το λόγο στον εισηγητή για συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω Εδώ μιλάμε για τις νομικές επιπτώσεις υφιστάμενων διατλαντικών συμφωνιών ε, για την προστασία, για την... Και αυτό φυσικά περιορίζεται σε αυτό. Οι διάφορες παρατηρήσεις ε, είναι συμπεράσματα γενικότερα για τη διαδικασία, όχι στα πλαίσια αυτής της έκθεσης αλλά ως ε, πολιτικές επιπτώσεις ε, που πρέπει να λαμβάνονται και αυτές υπόψη. Όμως ε, δεν είναι αυτό το πλαίσιο εδώ. Αυτό να το πω. Από την άλλη να πω ότι υπάρχουν και άλλες διμερείς συμφωνίες όπως αυτή στα πλαίσια της Europol. Εδώ υπάρχουν και η Ρωσία όμως ε, το να μιλάμε για διμερείς συμφωνίες σε 28 κράτη-μέλη, η Ρωσία, η Ευρωπόλ δεν είναι διμερείς. Ναι, αλλά είπατε ότι και θα έπρεπε να έχουν κάποια επιρροή και άλλες διμερείς συμφωνίες, αλλά εγώ θέλω να πω ότι εδώ δεν έχει να κάνει με τη Ρωσία, αλλά με την NSA είναι συγκεκριμένα πράγματα που δεν τα συμπεριλάβαμε. Θα μπορούσαμε να διευρύνουμε, αλλά δεν ήταν εδώ αυτό το καθήκον μας. Να πω γενικά ε, για την Safe Harbor. Να έχουμε πάντοτε ενώπιό μας πώς θέλουμε εμείς, όπως είπε η κυρία Ζέλα γενικά, πώς θέλουμε τα δεδομένα να φεύγουν από τη χώρα μας ή την Ήπειρό μας. έχουμε μια ρύθμιση που θα είναι σε έναν κανονισμό, σε μια οδηγία και θα διασφαλίζει ότι η μεταφορά των δεδομένων σε τρίτες χώρες θα πληρεί κάποια συγκεκριμένα στάνταρ προστασία δεδομένων. Αν καταγγείλουμε την Safe Harbor θα πρέπει να έχουμε μια άλλη βάση να βρούμε μια άλλη βάση για να έχουμε αυτά τα στάνταρ τα επαρκή για την προστασία. Είτε ονομάζεται Safe Harbor ή, οπωσδήποτε, ή έχει οποιοδήποτε άλλο όνομα. Χρειαζόμαστε όμως ένα κοινό στάνταρ για την ανταλλαγή δεδομένων γενικά χρειαζόμαστε φυσικά μια νομική βάση γι' αυτό. Όσον αφορά στο πρόγραμμα TFTP για το σύστημα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, να πω μια γενική παρατήρηση για τους ε, πολίτες. Έχουμε δύο βασικές μορφές μέτρων. Από τη μία έχουμε την παράνομη λήψη δεδομένων από ένα δίκτυο ή από ένα σερβερ και από την άλλη έχουμε την ζήτηση δεδομένων από μεγάλες εταιρείες οι οποίες κάνουν ανάλυση δεδομένων. Και στους δύο τομείς πρέπει στην ουσία, εντάξει, το παράνομο ε, μπορούμε να το λύσουμε πολιτικά, στον νόμιμο τρόπο θα πρέπει να θέσουμε στάνταρ, πρότυπα. Όταν μιλάμε για πάταξη της τρομοκρατίας ή της εγκληματικότητας και ταυτόχρονα για δεδομένα, θα πρέπει να αναρωτιόμαστε πώς θα ανταλλάσσουμε δεδομένα με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες για τις ε, τράπεζες δεδομένων, τα προγράμματα TFTP, το πρόγραμμα SWIFT, αν θεωρούμε λοιπόν ότι είναι σημαντικό να παρακολουθούνται τα, οι χρηματικές ροές της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας, θα πρέπει εμείς οι Ευρωπαίοι να είμαστε στη θέση να το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή το, κάνει, το κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε και γι' αυτό έχουμε μια συμφωνία με αυτούς. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σε καμία περίπτωση δεδομένα που να μας δείχνουν κάποιο χαρτί ας πούμε που να λέει ε, που να αναφέρει πώς γίνεται υποκλοπή δεδομένων. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή με δεδομένο ότι έγινε κάτι τέτοιο. Αυτά που λέγονται από την Europol, αυτά που λέγονται από την Κομισιόν, από την ε, κυβέρνηση τον είπα μας διασφαλίζουν ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να αφαιθούμε σε αυτούς, αλλά από την άλλη δεν έχουμε και πραγματικά γεγονότα που να μας λένε ότι μπορείτε να καταγγείλετε το σύστημα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Έτσι λοιπόν, εδώ στο Κοινοβούλιο, όταν δεν ξέρουμε πώς θα γίνεται η ανταλλαγή δεδομένων με τις ΗΠΑ, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Πώς θα θέλαμε να γίνει κάτι τέτοιο ταυτόχρονα προστατεύοντας τα προσωπικά δεδομένα και την εθνική ασφάλεια των κρατών. Πρέπει να βρούμε ε, ε, μια χρυσή τομή. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι σωστό να παραμείνει η συμφωνία γιατί έχουμε ε, και κάποια κοινά στάνταρ για την ε, επιτόπου παρακολούθηση και δεν θεωρώ ε, ποια θα... ότι υπάρχει κάποια εναλλακτική. Και δεν είναι εναλλακτική να μην μεταφέρονται δεδομένα για να, και να μην παρακολουθούνται οι χρηματικές ροές, η χρηματοδότηση της δημοκρατίας. Κυρία Μορφάη, γενικά εκφραστήκατε για τα συμπεράσματα αυτού του εγγράφου. Δεν το βλέπαμε έτσι ως τώρα. Δεν μιλάμε για πιο συγκεκριμένη παρακολούθηση των διαφόρων συμφωνιών. Εμείς θέλουμε στην τελική φάση της ε, εκθεσής μας να επικεντρωθούμε σε αυτό. Γιατί εδώ δεν είχε νόημα να συζητάμε αν υπάρχει παραβίαση ή όχι. Τελικά στην ουσία για το SWIFT και το TFTP δεν έχουμε πραγματικά γεγονότα στα χέρια μας που να μας λένε ότι κάποιος παρενέβη με τα δεδομένα της SWIFT. Το Έχουμε κάποια στοιχεία αλλά όχι αποδείξεις τέλος πάντων να το πω έτσι. Το έγγραφο εργασίας που έχετε εδώ είναι κάτι που το γράψαμε λίγο βιαστικά γιατί τελικά γιατί μας το είχαν ζητήσει για 5 Δεκεμβρίου και έπρεπε να το κάνουμε σήμερα. Ίσως δεν ήμουν και πολύ ξεκάθαρος λοιπόν για αυτό το λόγο στις επεξηγήσεις μου να πω ότι γενικά πρέπει να έχουμε δύο κατευθύνσεις. Από τη μία να κοιτάξουμε τις νομικές επιπτώσεις αυτών των διατλαντικών συμφωνιών, αλλά να έχουμε και μια πολιτική αξιολόγηση. Και αυτό είναι ακριβώς ε, το ερώτημα εδώ ποιος θα είναι ο ρόλος ε, του Κοινοβουλίου όσον αφορά στη διαφάνεια. Παίζει και αυτό ένα ρόλο στα συμπεράσματα που θα πρέπει να βγάλουμε γενικά για το έγγραφο, αλλά όχι για αυτό το κομμάτι του εγγράφου. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έτσι ολοκληρώνουμε την συνεδρίαση αυτή και μάλιστα 15 λεπτά νωρίτερα. Πολύ ωραία να σας ανακοινώσω ότι η επόμενη ακρόαση θα είναι την 5η 5 Δεκεμβρίου στις 3 με 6.30. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να τα πούμε και την 5η λοιπόν.